θα υπογράψω έξι ε, νομοθετήματα τα οποία έχουν εγκριθεί στα πλαίσια της διαδικασίας συναποφάσεως και θα τα βρείτε στα σημερινά πρακτικά. Το τελικό σχέδιο της ε, ημερησίας διατάξεως που